Vamos. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ευρωβουλευτές που είναι εδώ σήμερα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και θα ήθελα να σας ζητήσω λίγο υπομονή και κατανόηση, διότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες και σε περίπτωση που υπάρχουν τεχνικά προβλήματα θα πρέπει να μας το πείτε και θα έρθει σε επαφή μαζί σας ε, ε, τεχνικός με όποιο ευρωβουλευτή παρακολουθεί την ε, συγκεκριμένη συνεδρίαση μέσω βιντεοδιάσκεψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους για το προσωπικό που πρέπει να βρίσκεται στο Κοινοβούλιο για τη διαχείριση του συστήματος ή για τους βουλευτές που βρισκόμαστε εδώ. Ο χρόνος λοιπόν της συνεδρίασης χρειάστηκε να περιοριστεί στις δύο ώρες το μέγιστο για τους ίδιους λόγους, για να περιορίσουμε κινδύνους και στις καμπίνες των διερμηνέων, τους οποίους ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ. Ε, ο μέγιστος αριθμός των ε, γλωσσών σήμερα είναι έξι Αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά και γαλλικά. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης το απογευματινό ωράριο ακυρώθηκε και η Ολομέλεια ενέκρινε αρκετά κείμενα την προηγούμενη Πέμπτη. Σήμερα ε, πρόκειται να ψηφίσουμε δύο κείμενα, αλλά μας επιβεβαιώθηκε ότι η διάσκεψη των Προέδρων ε, των Επιτροπών δεν ενέκρινε ακόμα τις κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφοφορία στις επιτροπές. Ε, ε, είναι τα σημεία 4, 5 και 7 της ημερήσιας διάταξης. Επομένως, ε, πρέπει αυτές οι δύο ψηφοφορίες να αναβληθούν και όταν η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών θα μπορέσει να εγκρίνει τη διαδικασία ψηφοφορίας, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ψηφοφορίες εντός του Απριλίου. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις για την τροποποιημένη ημερήσια διάταξη, θεωρώ ότι εκρίνεται. Σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προεδρίας. Έχουμε το σημείο 2.1 που είναι η έγκριση των συστάσεων των συντονιστών βάσει του άρθρου 214 οι απαντήσεις ε, των συντονιστών των συνεδριάσεων από τις 19 και 20 Φεβρουαρίου του 2020, καθώς και τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας μετά από την ακύρωση της συνεδρίασης ε, της 17 η Μαρτίου του 2020. Ε, μπορείτε να τα βρείτε λοιπόν όλα αυτά στα έγγραφα της συνεδρίασης και να δείτε τις σχετικές απαντήσεις. Δεύτερον, ορισμός εισηγητών. Ο κύριος Ερικ Μαρκάρ από τους Πρασίνους ε, είναι εισηγητής της έκθεσης εφαρμογής ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για το άρθρο 43 της Οδηγίας ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τις κοινέ διαδικασίες, για την παραχώρηση και απόσυρση διεθνούς προστασίας. Ο Χουάν Φερνάντο Λόπε Αγγιλάρ είναι εισηγητή ε, του ψηφίσματο τη ΛΥΜΠΕ για τι υποχρεώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα αμοιβαιότητα των θεωρήσεων διαβατηρίων βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού. Και η κυρία Σύρα Ρέγο από την ΚΟΕ είναι εισηγήτρια για την γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ, για την έκθεση εφαρμογής της ΑΦΕ, της και της ΜΠΑΤΖ, για τα ε, πιστοτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Εάν η Επιτροπή εγκρίνει τις αποφάσεις και τις συστάσεις ε, των συντονιστών βάσει του άρθρου 214, ε, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Σημείο 3.3. Η έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. Πιο συγκεκριμένα, 14 Οκτωβρίου του 2019, 2 και 3 Δεκεμβρίου του 2019, 9 Ιανουαρίου του 2020 και 6 Φεβρουαρίου του 2020. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις για τα πρακτικά, εγκρίνονται και τα πρακτικά. Περνάμε τώρα στο σημείο 6. Η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης ε, στην Ελλάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από διάφορες ε, αναβολές, σήμερα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, για την κατάσταση στην Ελλάδα, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την προοπτική της μετανάστευσης και του ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τη διαχείριση των συνόρων. Έχουμε σήμερα ένα κατάλογο διακεκριμένων ομιλητών οι οποίοι θα συνδεθούν μαζί μας από διάφορες ε, μεριές ε, της Υπήρου μας. Θα έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την Ελλάδα, τον Νότι Μηταράκη από ε, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελλάδα, τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Αντιπρόεδρο για την Πρόωθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ήλβα Γιώχανσον, Επίτροπο για τις εσωτερικέ Υποθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Τερεσίγια Γκρά, από την Προεδρία του Συμβουλίου, ε, Υπουργό για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Υποθέσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Κροατίας, το Φαμπρίζες Λεζερή, ε, εκτελεστικό διευθυντή του Frontex και το Μάικελ Φλάχερτη, διευθυντή της Υπηρεσίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της ΦΡΑ. Ο στόχος αυτής της ανταλλαγής απόψεων είναι να μάθουμε τι μέτρα εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή ή τα οποία θα, τι μέτρα θα πρέπει να σχεδιαστούν για να συνεχίσουμε να βοηθούμε την Ελλάδα στην αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόλων και την υποδοχή των ετούντων άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και την αλληλεγγύη και την ε, ε, ισότιμη ε, κατανομή των ευθυνών, ταυτόχρονα εγγυόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων. Ελπίζουμε ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα αποτελέσει τη βάση των εργασιών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τη μελητική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, καθώς επίσης και τις ε, κατεπίγουσες ε, απαντήσεις σε νομοθετικό και μη νομοθετικό επίπεδο, σε επίπεδο ε, εισόδων σε πολύ μεγάλο αριθμό και υπάρχει πρόβλημα με τα διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε καλέσει και τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού να συμμετέχει εν ώψη και της πρότασης ε, που ενέκρινε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν διορθωτικό προϋπολογισμό για την επιπλέον χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ελλάδα. Θα παρέμβει ο αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής, ο κύριος Χέρβεστ, Όβερτβελτ. Ο χρόνο λοιπόν για τι ανταλλαγέ απόψεων είναι περιορισμένο. Θα δώσω λοιπόν καταρχά το λόγο στου ομιλητέ μα για 7 λεπτά τον καθένα και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο κύριος των παρεμβάσεων. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ο πρώτος. καλωσορίσατε Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Mr. Chrysokoidis, you have the floor. Κύριε Χρυσοχοίδη, έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Please press Thank the speak you. button. Oh, señor Chrysokoidis, puede usted hablar. Κύριε Χρυσοχοίδη, μήπως μπορείτε να μιλήσετε, είστε παρόν. Por favor, puede usted... Παρακαλώ, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να μπορέσετε να μιλήσετε. Πατήστε το κουμπί. Continúo con el siguiente. Okay. El siguiente. Okay. One minute. We're waiting for the connection. Περιμένουμε τη σύνδεση. Κύριε Χρυσοκοίδη, μήπως μπορείτε να πατήσετε το speak και να ξαναδοκιμάσετε να μιλήσετε. Si on doit continuer avec le reste de la liste indiqué. Oui, on continue. Avec les oui. Vamos a continuar con... Θα συνεχίσουμε με τον επόμενο μιλητή του καταλόγου, τον κύριο Μηταράκη. Κύριε Μηταράκη, είστε παρόν? Κύριε Μηταράκη. Έχετε το λόγο. Για 7 λεπτά. you push the Πατήστε το κουμπί, κύριε Μηταράκη. Who's working? I have to press, or they have to press. Press the button. Please push the button. Παρακαλώ, πατήστε το κουμπί για να μπορέσετε να μιλήσετε.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 Ε, please, the speak. Παρακαλώ, πατήστε το κουμπί speak για να μπορέσουμε να, ξεκιν... να σας ακούσουμε. And continue with Mrs. Okay. Mr. Skinas. Ο κύριος Σκινάς. Α, με ακούτε? Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί σας. Speak. Mr. Kinas. Κύριε Σχοινά, είστε εδώ. Με ακούτε. Oh. Can you hear me? <laughs> yes course. Thank ε, Ακούτε. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους. Το έχω υποσχεθεί, πάτησα όλα τα κατάλληλα κουμπιά από εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που είμαστε μαζί εικονικά. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Το έργο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων τις τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω απέδειξε την ανθεκτικότητά μας και την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει σε καιρούς κρίσης και την αποφασιστικότητά μας ε, να παραμείνουμε στην σωστή πορεία παρά το ότι έλεγαν ε, διάφοροι και έχουμε βέβαια ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με τη σημερινή συνεδρίαση. Να περάσω τώρα στο θέμα της σημερινής ημερησίας διάταξης. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ε, άνευ οι ηγέτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι ήταν ε, παρόντες σε ένα άλλο απτό και άνευ προηγουμένου δείγμα αλληλεγγύη στα εξωτερικά μας σύνορα τον Μάρτιο ξεκαθάρισαν ότι το καθήκον αυτό δεν μπορεί να το επομιστεί η Ελλάδα μόνη της. Είναι ευθύνη ολόκληρης της Ευρώπης και έχουμε δείξει πέραν πάσης αμφιβολίες ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν εξαιρετικές πιέσεις. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι το συνολικό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης που εγκρίναμε στις 4 Μαρτίου ήδη έχει αποτελέσματα. Οι δύο Ταχείες επιχειρήσεις στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα από την Frontex ε, ξεκίνησαν και είμαι σίγουρος ότι και ο Φαβέη ε, θα σας πει τα σχετικά. Μετά από την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από την Ελλάδα, τα κράτη-μέλη προσέφεραν 90.000 ε, αντικείμενα βοήθειας, βοήθεια η οποία χρειαζόταν ιδιαίτερος τις δύσκολες αυτές στιγμές. Και τέλος, οικονομική βοήθεια μέχρι του ποσού των 700 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί στην Ελλάδα 350 εκατομμύρια ευρώ άμεσα διαθέσιμα. Την προηγούμενη εβδομάδα προτείναμε τον τροποποιημένο προϋπολογισμό για τα επιπλέον 350 εκατομμύρια τα οποία θα ψηφίσει ε, προσεχώς η Επιτροπή σας. Θυμάμαι ακόμα υπό την προηγούμενη μου ιδιότητα πόσο γρήγορα μπόρεσε να ψηφίσει το 2015 τον τροποποιητικό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου για να τριπλασιάσει το ποσό των χρημάτων που είχαμε τότε στο πρώτο κύμα της κρίσης. Με την στήριξη λοιπόν της Frontex και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης έχουμε ένα νέο σχέδιο εθελοντικών επιστροφών που θα ξεκινήσει το στόμο των αλλά στηρίζουμε τις ελληνικές αρχές για να προωθήσουν την εθελοντική επιστροφή 5.000 ατόμων τα οποία έφτασαν ε, πριν από την 1η Ιανουαρίου στα νησιά για να υπάρξει μια αποσυμφόρηση εκεί πέρα και επίσης ε, θα έχουμε και επιπλέον ειδικού που θα στείλουμε στα, στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου που γνωρίζετε ότι είναι ήδη πάρα πολύ ταλαιπωρημένη στα όρια της ε, και βεβαίως η άμεση αυτή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την επομένη ε, του ξεσπάσματος της ε, κρίσης απέδειξε την ανθεκτικότητά μας και νομίζω θα το επιβεβαιώσουν και οι Υπουργοί ότι η κατάσταση στα σύνορα με την Τουρκία φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί αυτό το οποίο κάναμε τις τελευταίες τρεις-τέσσερις εβδομάδες απέδειξε σαφώς ότι κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει, να εκφοβίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δοκιμάζεται το σύστημά μας, ε, υπερισχύει ενότητα. Να έρθω τώρα στα σχέδιο ανάγκης της ε, Ελλάδας για τα ζητήματα του ιού, του COVID-19, που είναι επίσης μια δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί βεβαίως ε, ο αρμόδιος επίτροπος ε, τα έχει συζητήσει αυτά με, τον, με την η αρμόδια επιτροπός με τον Υπουργό τον κύριο Μηταράκη και άλλους οπότε θα σας ενημερώσει λεπτόμερος ε, όπως θα κάνει άλλωστε και για την πρωτοβουλία μας για την μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ελλάδα και ευχαριστώ τα κράτη-μέλη που ήδη έχουν ε, αναλάβει δέσμευση για να μας βοηθήσουν ως προς αυτό. Ε, τώρα θα αναφέρω και το ευρύτερο έργο μας ε, στο θέμα του κορονοϊού για ζητήματα εσωτερικών. Γνωρίζετε όλοι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ε, για να περιοριστούν τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα μήνα. Η κατάσταση νομίζω μας αναγκάζει να ανανεώσουμε αυτούς τους περιορισμούς υπό συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ε, που εκδώσαμε αυτήν την εβδομάδα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε άλλωστε. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα που έλαβαν ουσιαστικά όλα τα κράτη-μέλη στα εσωτερικά μας σύνορα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια εξαιρετική κατάσταση η οποία δικαιολογεί αυτές τις αποφάσεις, αλλά θέλουμε αυτό να γίνει έφτακτα, σύμφωνα με τις καθημερινές γραμμές που έχουμε καταρτήσει με τα κράτη-μέλη και θέλουμε να υπάρξει και ένας ορίζοντας ε, που θα επιτρέψει να επανέλθει η κατάσταση στο κανονικό. Να καταλήξω λοιπόν κυρία Πρόεδρε λέγοντας ότι όσο συμβαίνουν όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο διαχείριση κρίσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δουλειά μας δεν θα πρέπει να είναι μόνο διαχείριση κρίσης. Κομμάτι της αντιμετώπισης της κρίσης είναι το να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρούμε σε όλες τις πτυχές της εργασίας μας και δεν θα αποσταθεροποιηθεί το σύστημα. Και τις δύσκολες αυτές ώρες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε παράλληλα, όχι μόνο στα άμεσα, τα τρέχοντα, αλλά και σε μεσομακροπρόθεσμες δράσεις αφενός για να στηρίξουμε την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των εξαιρετικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει συμμορφούμενοι πλήρω με το ευρωπαϊκό δίκαιο, θεμελιώδη δικαιώματα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και από την άλλη να συνεχίσουμε την εντατική μας εργασία για να προτείνουμε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο για το οποίο εγώ και η κυρία Γιώχανσον έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή. Θα ήθελα λοιπόν να αποστείλω αυτό το μήνυμα, αυτή την διαβεβαίωση ότι η δουλειά μας συνεχίζεται και είναι επίσης σαφές ότι θα λάβουμε υπόψη ε, στη δουλειά που κάνουμε τις εξαιρετικές συνθήκες ε, που ήταν απρόβλεπτες αλλά ε, αντιμετωπίζουμε τώρα όσον αφορά την πανδημία του COVID-19. Θα συνεχίσουμε να ζητούμε βιώσιμες λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για αυτήν την συζήτηση σήμερα εσάς και τον κύριο Λόπεζ Αγγιλάρ, τον οποίον είδα πιο πριν ε, ψηφιακά και διαβεβαιώ και εσάς και όλους τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων με τους οποίους είμαστε σε στενή επαφή ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ανεφροηγούμενη κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρία Γιωχάνσον, Κυρία Επίτροπε, μας ακούτε? Πιέσατε παρακαλώ. Το κομβίον. Μ' ακούτε? No connection. We continue. Δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίζουμε. Α, κι όμως. Έχετε τον λόγο. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης και κατά πάσα πιθανότητα θα χειροτερεύσουν τα πράγματα πριν να αρχίσουν να βελτιώνονται. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε σε καιρό κρίσης είναι άμεσες επιχειρησιακές δράσεις Δεύτερον, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών μελών και παγκοσμίω είναι η κατάλληλη στιγμή να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και να προστατεύσουμε και την ικανότητα να βοηθήσουμε. Και τρίτον, σε καιρό κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρήσουμε τις αξίες μας και να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε κρίση, όχι μόνο η κρίση για τον κορονοϊό, αλλά η οποιαδήποτε άλλη κρίση, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευση του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καταβληθμοί προσφύγων ε, δεν είναι εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουν το μεγάλο αριθμό ατόπων που ζουν σε επισφαλές συνθήκες και αν υπάρξει εξάπλωση του ιού και μπορεί να υπάρξει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι επικίνδυνο και για τους πρόσφυγες που βρίσκονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτούς που ζουν σε απα... Ε, απαράδεκτες συνθήκες στα ελληνικά νησιά. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ελλάδα είχαμε κάποιες πρώτες ε, περιπτώσεις, ένα καταβλισμό προσφύγων εκτός ε, Αθηνών. Έχουμε 20 επιβεβαιόμενες ε, περιπτώσεις εκεί. Νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμο, είναι ένα ε, καταβλισμός στον οποίο υπάρχει πολύ καλή διαχείριση και υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά φυσικά κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου. Ε, έχουμε και κάποια περιστατικά στη Λέσβο, εκτός όμως των καταβλισμών των μεταναστών και των προσφύγων. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αναλάβουμε αμέσω δράση για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές αρχές βεβαίως είναι υπεύθυνε, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τεράστια υποστήριξη και θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε όμως και τεράστια υποστήριξη και από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ε, Είμαστε σε μόνιμες σχεδόν επαφές με την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές και αποφασίσαμε για ένα σχέδιο δράσης κατεπίγουσας απάντησης. Δεν θα σας αναφέρω όλο το σχέδιο, αλλά περιλαμβάνει για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσει με την κατάσταση των πιο ευάλωτων εκτός ε, των ε, ε, καταβλισμών σε ε, δωμάτια ξενοδοχείων τα οποία είναι προετοιμασμένα και είναι αυτή τη στιγμή κενά, ώστε να μην υπάρξει ε, μετάδοση όταν και εφόσον, ε, εάν φυσικά, ε, ο ιός φτάσει στους καταβλισμούς. Πρέπει επίσης να ε, υπάρξει και ιατρική υποστήριξη και στα νησιά και για τους μετανάστες, αλλά και φυσικά και για τον πληθυσμό των νησιών. Έχουμε ήδη υποστήριξη με ιατρικό εξοπλισμό και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη. Θα πρέπει οι νέε αφήξει να είναι ξεχωριστέ από αυτού που βρίσκονται ήδη στον καταβλισμό. Θα πρέπει επίση να γίνονται δοκιμέ, τεστ και να φροντίσουμε αυτοί που είναι θετικοί στον ιό να ε, μπαίνουν αμέσως σε καραντίνα. Χρειαζόμαστε φυσικά και ε, περιορισμούς ε, στα ταξίδια και πρέπει να δίνονται και πληροφορίες για το τι θα πρέπει να γίνεται. Ε, αλλά ε, θα πρέπει να ε, μειώσουμε και τις πιέσεις στους καταβλισμούς αυτούς. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε τη μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουμε 8 κράτη-μέλη που δεσμεύτηκαν να υποδεχθούν 1.600 ασυνόδευτους ανήλικους και νομίζω ότι η πρώτη μετεγκατάσταση θα γίνει εντός αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη εβδομάδα πριν το Πάσχα δηλαδή και εργαζόμαστε σε πολύ θετικό πνεύμα με τα κράτη-μέλη αυτά που δείχνουν συγκεκριμένη αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Γνωρίζω ότι οι ελληνικές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι περίπου 2.000 ασυνόδευτοι ενήλικοι ε, είναι έτοιμοι για μετεγκατάσταση, έχει γίνει αξιολόγηση της ηλικία τους και έχουν και την σχετική τεκμηρίαση για να φύγουν. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα ήδη σε εξέλιξη για βοήθεια και παρέχεται φυσικά και πολύ χρηματοοικονομική στήριξη. Θα σας τα πω εντάχει υπάρχει αμέσως διαθέσιμα 350 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι υποστήριξη για ε, δυνατότητες υποδοχής στην ενδοχώρα, ε, ενοικίαση ε, στέγασης, επίδομα στους ε, μετανάστες και πρόσφυγες, περίπου 100 εκατομμύρια είναι όλα αυτά, υποστήριξη της δυνατότητας υποδοχής στην ενδοχώρα, 31 καταβλισμοί και διαχείριση που παρέχονται από τον ION, ε, περίπου 100 εκατομμύρια και αυτό, συνέχεια της στοχευμένης στήριξης για τη βασική προστασία για τις οικογένειες και τα παιδιά, ε, παροχή υπηρεσιών στην περιοχή του Καράτεπέ στη Λέσβο, την οποία διαχειρίζεται, η Πατιαρμοστία για τις πρόσφυγες, περίπου 25 εκατομμύρια, για τα, ε, πρόγραμμα προσωρινή στέγαση σε ξενοδοχεία για τα ευάλωτα άτομα τα οποία θα πρέπει να φύγουν από του καταβλισμού, περίπου 35 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα είναι ήδη διαθέσιμα και έχουν αρχίσει να ε, διατίθενται. Επίσης, έχουμε επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν για ε, του εξής σκοπούς. 280 εκατομμύρια θα διατεθούν για την κατασκευή πέντε νέων ε, χώρων υποδοχής και ταυτοποίησης ε, στα ελληνικά νησιά εντός του έτους για να υπάρχουν κατάλληλες δυνατότητες υποδοχής βάση και προτύπων. Η διαδικασία εθελοντικών επιστροφών και επανένταξης είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και στη συνέχεια οι υπηρεσίε στα νέου ε, στους νέους χώρους υποδοχής, μεταφορά τροφίμων, επιπλέον προσωπικό, οι ιατρικές ομάδες, καθώς επίσης και προηγμένη υποστήριξη στι υπηρεσίε ασύλου της Ελλάδος, 50 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, 50 εκατομμύρια προτείνονται να διατεθούν για ε, τα σύνορα και τις θεωρήσεις διαβατηρίων για να καλύπτεται το στόχο της ανάπτυξης ε, συνοριοφυλάκων και αστυνομικών ε, στα εξωτερικά σύνορα της, Ευρωπαϊκής, της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, 50 εκατομμύρια λοιπόν εκεί και επιπλέον προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες της Frontex η οποία θα ενισχυθεί με 10 εκατομμύρια ευρώ και τέλος 10 εκατομμύρια ευρώ στην ΕΑΣΟ για την αποστολή εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα. Επομένως, αυτά τα οποία ε, σας είπα ε, συμπληρώνονται με το εξή που είναι εξίσου σημαντικό αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου και καλωσορίζουμε την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που μου είπε ότι πλέον οι νέε αφήξει ε, του Μαρτίου θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τι αρχέ και τα θεμελιώδη δικαιώματά μα και τι αξίε μα, όπω είπα στην αρχή. Και αξιότιμα μέλη θα ήθελα να προσθέσω και το εξή. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει αυτό σε καιρό κρίσης ε, είναι πάντα κίνδυνος ε, να υπάρξει αύξηση της ε, ξενοφοβίας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την πολύ σημαντική συμβολή που έχουν δώσει άτομα τα οποία είναι μετανάστες, γιατροί που παρέχουν υπηρεσίες ή κάνουν θελοντική εργασία. Σε όλη την Ευρώπη οι μετανάστες κινητοποιούνται για να υποστηρίξουν τις χώρες που τους φιλοξενούν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και τέλος, καλωσορίζω τα μέτρα τα οποία οποία λαμβάνουν 7 κράτη-μέλη και περιοχέ για να διευκολύνουν πρόσβαση σε πρόσβιαση και υπηρεσίε υγεία, για μετανάστες και πρόσφυγε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να εφαρμόσουμε τι συστάσεις του ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία και να εξασφαλίσουμε ότι κανένα τομέα τη κοινωνία μα δεν θα μείνει πίσω και θα υπάρξει υποστήριξη για όλου. Θα ήθελα να τονίσω και τη σημασία του να υπάρχει μια κοινωνία που θα είναι πιο φιλόξενη. Ε, πολλοί μετανάστε βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση στη χώρα του, σε ευάλωτη κατάσταση στην αγορά εργασία, τεράστιο κίνδυνο για ανεργία ε, και ε, για οικονομικού πόρου. Για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και του ρατσισμού και για να βοηθήσουμε τους ευάλωτους μετανάστες, θα ε, κάνω μια διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, ε, τα συνδικάτα και τους εργοδότες για να μπορέσουμε να δούμε επιλογές για την προστασία και την υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων και την ε, μεγιστοποίηση της συμβολής τους ε, στην φάση της ανάκαμψης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Γκράς είναι εδώ. Κυρία Γκράς. Με ακούτε? Push the button. Πατήστε το κουμπί. Talk. Hello, can you okay. hear me? Okay. Welcome. Welcome. You have the floor, have the floor. for seven thank minutes. You. Seven minutes. And thank you. And thank you. Thank you, Mrs. Chair. Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές και επίτροποι. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, που συγκάλεσε την βιντεοδιάσκεψη αυτή για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα. Ε, δείχνει την σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό και σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες. Μετά την ανακοίνωση των τουρκικών αρχών ότι ανοίγουν τα σύνορα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο αντέδρασε άμεσα δείχνοντας ε, συγκεκριμένη απτή αλληλεγγύη προς ε, την Ελλάδα. Και όλα τα κράτη-μέλη είπαν ότι είναι αποφασισμένα να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά στενά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα γίνουν ανεκτές παράνομες διαβάσεις των συνόρων. Σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αναγνωρίζουμε με την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζει η Τουρκία, απορρίπτουμε όμως ε, την χρήση ε, της πίεσης αυτής από την Τουρκία για πολιτικούς ε, σκοπούς και αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της δήλωσης του 2016. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεχίσει να στηρίζει τις κοινότητες των προσφύγων στην ε, Τουρκία, όπως ε, ε, έκανε και τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την απτή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, όλα τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν την στήριξή τους με διάφορα μέσα. Η Frontex ανταποκρίθηκε αμέσως ε, με την άμεση αποστολή δύο ομάδων Rabbit ε, κάτι το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα της Ελλάδος επίσης. Αποτέλεσε ένα σαφές μήνυμα της κοινοτικής αλληλεγγύης ε, και ένα αποτρεπτικό μέσο κατά αυτής της υποκινούμενης ε, πίεσης. Αυτά τα μέτρα πρέπει να συνεχιστούν για όσο απαιτείται και θεωρούνται απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο των περιορισμών που μας επιβάλλει ε, ο ιός η αποστολή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σύλλου άλλων 160 ειδικών στην Ελλάδα. Προχωράμε επιταχυμένη διαδικασία. Ήδη 40 άτομα έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί και μέχρι το τέλος Αυγούστου θα είναι όλοι οι επιχειρησιακοί. Επίσης η Ελλάδα ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας για εξοπλισμό για να καλυφθούν βασικές ανάγκες των ε, μεταναστών οι οποίοι φτάνουν. Τα κράτη-μέλη κινήθηκαν γρήγορα, η παράδοση των υλικών παρά τις περιπλοκές στα σύνορα ήταν επιτυχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε άμεση βοήθεια 350 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, ε, η οποία είναι διαθέσιμη για την διαχείριση των σύνορων και της μετανάστευσης. Τα περισσότερα έργα έχουν ήδη ε, δημοπρατηθεί όπως είπε και η Επίτροπος Γιώχανσον. Επίσης προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση σε σχέση με τον κορονοϊό στον πληθυσμό των μεταναστών. Ανέφερε επίσης ε, και τον ε, σχετικό σχεδιασμό η κυρία Γιώχανσον ως προς αυτό. Πολλά κράτη-μέλη είπαν πως είναι διατεθειμένα να μετακινήσουν, να συνοδευτούν ανηλίκους από την Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν γύρω στα 5.000 άτομα στην χώρα, 2.100 εκ των οποίων μπορούν να μετακινηθούν αμέσως. Είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές και τις υπηρεσίες της Κομισιόν για να υπάρξει αυτή η ανακατανομή. Όλες αυτές οι δράσεις είναι έκφραση της αλληλεγγύης μας με την Ελλάδα και δείχνουν ότι είμαστε ενωμένοι στην δέσμευσή μας για να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παρά κάποια περιστατικά μπορούμε να πούμε πως η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι σταθερή στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και να διασφαλίσουμε έναν συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων μέσω των σχετικών διάβλων. Τη Προεδρία την προηγούμενη εβδομάδα οργάνωσε μια ανταλλαγή πληροφοριών για να δούμε την κατάσταση στην διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ακολουθήσει άλλη μια ανταλλαγή πληροφοριών την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, η Προεδρία θα συνεχίσει την συνεργασία με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Καταλήγοντας, να σας ευχαριστήσω και πάλι που οργανώσατε αυτήν την βιντεοδιάσκεψη. Οι ιδέες που προκύπτουν από αυτές τις συζητήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για να βρούμε αποτελεσματικές απαντήσεις στις προκλήσεις ε, που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Χρυσοχοίδη, με ακούτε? Πάτησε το κουμπί. Welcome, you have the floor. Welcome, you have... Καλώς όρισατε, έχετε το λόγο, έχετε 7 λεπτά. Push the button, please. Παρακαλώ πατήστε το κουμπί. Yes. Thank you. Welcome. Okay. Good morning. Good morning. Καλημέρα σας. Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα σε όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά στο τελευταίο εξάμεινο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και καταρχάς ε, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσία μου εδώ σήμερα μαζί σας και την δυνατότητα που μου δίνεται να παρουσιάσω τη θέση της χώρας μου για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι αυτονόητο φυσικά ότι η Ελλάδα ως ε, εξωτερικό κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, που ταυτόχρονα φυσικά είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσω λέγοντας ε, δύο λόγια για τα εξωτερικά μας σύνορα με την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία. Η κατάσταση με τις χώρες αυτές είναι πάρα πολύ καλή και δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η συνεργασία είναι καλή, είναι ε, καθορισμένη η διάβλη και τα δυνητικά προβλήματα αντιμετωπίζονται αμέσως και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, ε, το τελευταίο διάστημα, ενώ αντιμετωπίζουμε την πανδημία, και έχουμε φυσικά και τις γνωστές ε, ε, περιοριστικές διαδικασίες μετακίνησης. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα και ό,τι θέμα προκύψει αντιμετωπίζεται εγκαίρος και καταλήλως. Το βασικό σημείο ανησυχία για μας είναι τα σύνορά μας με την Τουρκία. Δεν θα ε, επαναλάβω τις πρόσφατες εξελίξεις επί του θέματος. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε όλοι τι συνέβη τον τελευταίο μήνα και το μόνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η μαζική κίνηση μεταναστών δεν ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, ήταν μια χειραγώγηση κατόπιν προτροπής των τουρκικών αρχών. Η αντίδραση της Ελλάδος ήταν ε, η κατάλληλη και έγινε γέρος ε, σε επιχειρησιακό επίπεδο και καταφέραμε επιτυχώς να προλάβουμε την ε, σημαντική σρωή μεταναστών οι οποίοι συγκεντρώνονταν σε μεγάλες ομάδες στα σύνορα ε, του ποταμού Εύρου και παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να προκαλέσουν ε, ζημίες ε, στο φράχτη, σε καθημερινό η βάση γινόταν κάτι τέτοιο, οι συνοριακές αρχές μας το αντιμετώπισαν διότι πολλές φορές πετούσαν πέτρες, δακρυγόνα και άλλα. Εμείς παραμείναμε αποφασισμένοι, ήρεμοι και με αποφασιστικότητα προστατεύσαμε τα δικά μας και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να διαβιβάσω και προς εσάς. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, διότι για μας αυτό είναι ζωτική σημασία πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα. Και θα ήθελα να σας αναφέρω εδώ και κάποια άλλα θέματα ε, της παρούσας μεταναστευτικής κρίσης. Ένα από αυτά έχει να κάνει με το προφίλ των ατόμων που προσπαθούν ε, να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι ακούστηκαν κάτι άλλε ε, φήμες, η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων, περίπου το 70% είναι Αφγανοί, επίσης Πακιστανοί, νέοι άνδρες και κυρίως δεν έρχονται από τα μέτωπα του πολέμου, από το Ιντλίμπ στη Συρία, όπως ε, διέδιδαν ε, ε, οι τουρκικές πλευρές, αλλά, και εδώ έρχομαι και στο δεύτερο σχόλιο μου, για τη δημοσίευση και διάδοση ψευδών ειδήσεων, fake news από τις τουρκικές αρχές. Είναι λυπηρό αυτό το οποίο συνέβη και αναπαράχθηκε μάλιστα και από ε, κάποια μέσα ενημέρωσης ε, παγκοσμίως. Θα ήθελα εδώ ε, να τονίσω ότι παρά το γεγονός ότι υποστήκαμε βία η επίθεση, οι δυνάμεις μας έδρασαν επαγγελματικά, σεβόμενες πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ε, δικαιώματα. Κάτι το οποίο δεν έκαναν οι γειτονέ μας. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με το πνεύμα της αλληλεγγύης αποδείχθηκε ε, στη διάρκεια της κρίσης που αντιμετωπίσαμε η άμεση αντίδραση της Frontex και η άμεση ε, ανάπτυξη των επιχειρήσεων ε, Rapid και της πολύτιμης επιχειρησιακής υποστήριξης πολλών κρατών μελών ήταν αξιοσημείωτες πραγματικά και θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη εκτίμησή μας ε, και φυσικά να ευχαριστήσουμε. Εμείς ε, προσωπικά εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Σχοινά, την κυρία Γιώχανσον, την Επίτροπο και φυσικά και τον επικεφαλής του Frontex, ε, τον κύριο Φαμπρίς Λεζερή, ο οποίος ε, ήταν πάρα πολύ κοντά μας καθημερινά. Αντίστοιχα με ό,τι συνέβη στην περιοχή του Εύρου, αντιμετωπίσαμε ε, αντίστοιχα προβλήματα και στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Η τουρκική εκτοφυλακή, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, ήταν παντελώς απούσα και απέφυγε να απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα των ελληνικών εκτοφυλακών ε, για την πρόληψη της αναχώρησης μεταναστών από την άλλη πλευρά, από την τουρκική εκτογραμμή. Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην πανδημία την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά ε, στην εποχή μας, ε, στη γενιά μας, ε, που όλοι μαζί, όλα τα κράτη-μέλη, αντιμετωπίζουμε ένα κοινό εχθρό. Έναν εχθρό ο οποίος είναι ισχυρός, απρόβλεπτος και το πιο σημαντικό είναι αόρατος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι ενωμένοι για να υποστηρίξουμε ένα τον άλλον και ιδίω ε, τα κράτη-μέλη που πλήττονται περισσότερο. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη, την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη και όταν ε, περάσει η κρίση να είμαστε πιο δυνατοί σοφότεροι και να επιβεβαιώσουμε τις κοινέ μας ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Χρυσοχοίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον Υπουργό κύριο Μηταράκη. Με ακούτε? Please, push the button. Παρακαλώ πιέστε το κουμπί. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο. Για 7 λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιμετωπίζουμε μια μεταναστευτική κρίση με αυξημένες ε, αφήξεις από τον περασμένο Ιούλιο. Σας τα είπε και ο κύριος ε, Χρυσοχοίδης. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις δυνατότητες υποδοχής, αντιμετωπίζουμε τεράστιες ε, πιέσεις. Έχουμε 100.000 άτομα σε κέντρα ή σε στέγαση, εκ των οποίων 40.000 είναι στα νησιά και 19.000 ε, στην ε, Μόρια. Υπάρχουν τρεις λόγους. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τον οποίο να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είχαμε μία αύξηση 86% των αφήξεων από τον Ιούλιο του 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ε, έχουμε μία αργή διαδικασία αποφάσεων και τρίτον λόγω των περιορισμών της κοινή δήλωσης ε, με την Τουρκία που δέχεται επιστροφές μόνο από τα νησιά, έχουμε περιορισμένες ε, μετακινήσεις από τα νησιά στην ε, υπηρετική χώρα. Παρά αυτούς τους περιορισμούς, το πρώτο εξάμεινο του 2020, 10.000 άτομα μεταφέρθηκαν στην υπηρετική χώρα. Συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν, με την Ήλβα και το Μαργαρίτη για να αυξηθεί ο αριθμός αυτό στο δεύτερο εξάμεινο και έχουμε και το πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών για 5.000 άτομα που ανακοινώσαμε πρόσφατα με την κυρία Γιώχανσον. Για να βελτιωθούν οι συνθήκες και να αυξηθούν οι δυνατότητες χρειαζόμαστε αυτή την χρηματοδότηση για τα νέα κέντρα υποδοχής στα νησιά για να αντικατασταθούν η Μόρια, το Βιάλ και το Βαθύ. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη Μόρια σε μια μέρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε σοβαρές αλλαγές μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στην υπηρετική χώρα. Έχουν δύο ήδη ολοκληρωθεί, στη Μαλακάσα και τις Σέρες και θα μεταφέρουμε 2.000 άτομα από τα νησιά. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις σε διαμερίσματα. Έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση για 5.000 επιπλέον θέσεις και συνεργαζόμαστε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για 10 με 15.000 επιπλέον θέσει. Ε, πρέπει να οριστικοποιηθεί αυτή η χρηματοδότηση επιγόντω. και επίσης πρέπει να επιβάλλουμε την κοινή δήλωση όπως ανέφερε και η Προεδρία και να τροποποιηθεί έτσι ώστε να μειώνει τις ροές, να επιτρέπει τις ε, επιστροφές ατόμων που, των οποίων η έτσι έχει απορριφθεί να μην αφορά τα άτομα που είναι μόνο στα νησιά για να μην υπάρχει ακριβώς αυτός ο συνοστισμός ε, στα νησιά και να παρέχει και ένα ρόλο στη Frontex. Επίση ε, πρέπει να πούμε πως ε, η Τουρκία μας ειδοποίησε ότι δεν δέχεται επιστροφές λόγω COVID. Μιλώντας για τον ιό, από την αρχή της κρίσης είχαμε γύρω στα 1500 κρούσματα, 51 νεκρούς συνολικά, έναν χτες και έναν σήμερα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο στην υπηρετική χώρα, καθώς τα νησιά είναι πιο προστατευμένα. Επίσης, σήμερα δεν είχαμε κρούσματα στα κέντρα υποδοχής στα νησιά. Ένα, μία εγκατάσταση μόνο επηρεάζεται στην υπηρετική χώρα, πολύ κοντά στην Αθήνα. 20 άτομα είναι θετικά, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και για να περιοριστεί και η κίνηση επίσης από τα στρατόπεδα αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν για την κατάσταση στα νησιά και τις συμμερίζομαι και εγώ αυτές τις ανησυχίες. Εργαζόμαστε σκληρά και έχουμε λάβει μέτρα τα οποία είναι τα εξή. Πρώτα απ' όλα από 1η Μαρτίου ε, διαχωρίζουμε τις νέες αφήξεις. Ε, οι νέες αφήξεις δεν πάνε στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Περιορίζουμε επίσης την πρόσβαση από και προς τις εγκαταστάσεις. Φτιάχνουμε ειδικέ εγκαταστάσεις υγειονομικές εντός των δομών και ενημερώνουμε επίσης και τους κατοίκους στην γλώσσα τους ε, για τα θέματα του COVID. Είναι σαφές ότι το σύστημα υγείας ε, αντιμετωπίζει πίεση, οι πόροι δεν είναι άπειροι. Συνεργαζόμαστε στενά με την ε, Κομισιόν, την Υπατερμοστία του ΟΗΕ, τον Ερθρό Σταυρό, τον Διεθνή Οργανισμό μετανάστευση για τους χωρί σύνορα και άλλους. Κάποιοι είπαν ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε τα άτομα στην υπηρετική χώρα ε, δηλαδή από περιοχές οι οποίες ε, δεν έχουν κρούσματα σε περιοχές που έχουν κρούσματα. Δεν υπάρχουν θέσεις όμως, θα απαιτηθούν περαιτέρω κονδύλια για περαιτέρω θέσεις, αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε λίγες μέρες. Οποιαδήποτε επίση προσφορά με την κατάσταση στα κράτη-μέλη είναι ευπρόσδεκτη γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση μόνοι μα. Ε, προσωπικά εγώ ζω στην Χίο και γνωρίζω το πρόβλημα από πρώτο χέρι. Για το θέμα του ασύλου βελτιώνουμε το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να και ποιοτικέ αποφάσει σεβόμενοι πλήρω τι διεθνεί μα υποχρεώσεις ε, σε συντομότερο χρονικό διάστημα κατόπιν είναι σημαντικό για να μην μένει ο κόσμο στις δομές υποδοχής και έχουμε πάρα πολύ στήριξη από την ΕΑΖΟ. Πάγωσαν οι αιτήσει τον Μάρτιο δεδομένη της κατάσταση στα σύνορά μα. Ε, εκτιμούμε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχήσεις, ε, τι οποίες εξέφρασε και η Ήλβα. Λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα δεδομένων των συνθήκων. Υπήρχε νομική βάση για αυτήν την απόφαση. Έπρεπε να προστατεύσουμε την εθνική μα ασφάλεια, δημόσια τάξη και δημόσια υγεία. Δεν ε, υπάρχει πλέον αυτό το πάγωμα. Από 1η Απριλίου επανήλθαμε στην κανονική διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω με το εξή. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εξακολουθούν να είναι ο πιο ευπαθής πληθυσμό. Αναζητούμε μια λύση για να μεταφερθούν όλοι από τα νησιά ε, πρώτα απ' όλα σε κέντρα διαλογής, να δούμε ποιοι ε, δικαιούνται προστασία, και μετά οι υπόλοιποι να μεταφερθούν σε κέντρα κατάλληλα για την ηλικία του τέλο. οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πάνε σε κέντρα στην υπηρετική χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Κομισιόν, ειδικά την κυρία Γιώχανσον και τα κράτη-μέλη για τι πρωτοβουλίε με την κατάστασή ανηλίκων, ειδικά τα κράτη-μέλη τα οποία προσφέρθηκαν ε, για μετεγκατάσταση αυτές πολύ δύσκολες μέρες με την κρίση του κορονοϊού. Τέλος, και τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος ε, ήταν πρώην Ευρωβουλευτής και συντονίζει μια διάσκεψη για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λετζέρη, με ακούτε? Πατήστε το κουμπάκι παρακαλώ. Κύριο Φλάχερτη, με ακούτε. Κύριε Λετζέρη, εσείς, με ακούει κάποιος. Μιλήστε παρακαλώ, πατήστε το κουμπί. Όχι. Κύριο Φλάχερτη. Με ναι, ακούτε, μπορείτε να μιλήσετε. Ακούσουμε τον κύριο Χέραπς. Α, ο κύριος Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την πρόσκληση για να συμμετέχει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που είχε μεγάλη ε, επαφή με την κατάσταση στην Ελλάδα από το 2017 και ήμουνα κι εγώ πριν από δύο εβδομάδες εκεί. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ισχυρή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, καθώς επίσης και με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες. Πριν περάσω σε συγκεκριμένα σημεία, θα ήθελα να αναφέρω δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμη λύση διότι η κατάσταση που συζητούμε σήμερα χωρίς ε, αλληλεγγύη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Και δεύτερον, όταν αναφερόμαστε σε θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό, αναφερόμαστε στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των μεταναστών αλλά και του τοπικού πληθυσμού, όπως για παράδειγμα του πληθυσμού των νησιών. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα του COVID-19 και των ε, καταβλισμών προφύγων, ο ο οξύς κίνδυνος έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Εκτιμούμε τις δράσεις των ελληνικών αρχών τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου να εξασφαλίσουμε και απόσταση μεταξύ των ίδιων των μεταναστών. Για παράδειγμα, όπως ε, ανέφερε και η Επίτροπος ε, Γιώχανσον, να χρησιμοποιούνται ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στα νησιά, ώστε να υπάρχει και ε, απόσταση. Επίσης, θα θέλαμε να υπάρχουν και δυνατότητες απολύμανσης σε μεγαλύτερο βαθμό στους καταβλισμούς και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν τις ε, διαδικασίες αλσίλου ε, και ε, για τις εγκαταστάσεις αυτές και παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε η σε αυτή τη στιγμή αλλά θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε και πάλι εικονικά εργαλεία. Χρησιμοποιήθηκε το Skype με ανάμεικτα αποτελέσματα αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα προβλήματα είναι ασήμαντα. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα των καθυστερήσεων των διαδικασιών ασύλου, αυτό δημιουργεί θέματα προθεσμών και για την επανένωση ε, των οικογενειών και προτρέπουμε και άλλα κράτη-μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν τις ε, προθεσμίες ε, δεδομένων των συνθήκων. Επειδή υπάρχει ε, υπερπληθυσμός ε, στους καταβλισμούς, ε, είναι ευπρόσδεκτες οι πρωτοβουλίες για την επανεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Υπήρχε και ένα σημείωμα για υποστήριξη των κρατών μελών που θα υποδεχθούν αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά και θα υπάρξει και έκθεση και θα δούμε τις καλές πρακτικές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τις επόμενες εβδομάδες. Ένα βασικό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό σήμερα είναι να αποφύγουμε να επιλέγουμε παιδιά ανάλογα με κριτήρια τα οποία δεν υποστηρίζουν κανένα κοινωνικό σκοπό, όπω για παράδειγμα την εθνικότητά του, ε, την ημερομηνία άφηξη στην Ευρώπη ή την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν τα παιδιά αυτά. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα των αφήξεων του Μαρτίου, ε, καλωσορίζουμε την απόφαση να μην συνεχιστεί η αναστολή της διαδικασίας ασύλου, αλλά μας ανησυχεί η μοίρα αυτών που έφτασαν στη διάρκεια του Μαρτίου. Θα θέλαμε να προτείνουμε οι ελληνικές αρχές να εφαρμόσουν αναδρομικά τη διαδικασία ασύλου για το Μάρτιο και να υπάρχει και έγκαιρη πρόσβαση στις διαδικασίες αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους. Και Κατά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου θα θέλαμε να εργαστούν σε αξιοπρεπείς ε, εγκαταστάσεις. Επίσης, εκφράζουμε και την ανησυχία μας όσον αφορά την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, διότι ε, μπορεί κάποιοι να ε, έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας και αν εκκρεμούν ε, ε κυρώσεις από αυτών, μπορεί να υπάρχει θέμα ε, διεθνούς δικαίου. Και τέλος θα θέλαμε να ζητήσουμε από τις αρχές στην Ελλάδα να φροντίσουν να μην υπάρχει καμία παράνομη επιστροφή αυτών που έφτασαν στη διάρκεια του μηνό ε, Μαρτίου που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ε, επαναπροώθησης. Και τέλος θα ήθελα να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε εκφράζοντας την εκτίμησή μου για τις αδελφές Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με τη Frontex για να εφαρμόσουμε ε, δυνατότητες παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα διαδραματίσουν φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο δεδομένων των συνθηκών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Φλάχερτη. Και τώρα ο κύριος Λεζερή. Ε, μ' ακούτε κύριε Λεζερή. Ο κύριος Λεζερή. Μπορείτε να μιλήσετε, να πατήσετε το κουμπί. Mr. Legeri, can you... Κύριε Λεζερή, με ακούτε? We're waiting for a minute. Μένουμε ένα λεπτό. Probably we... we can talk. Okay. Okay. Okay. We're waiting, but we continue. Περιμένουμε, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συντονιστές. Υπάρχει φυσικά πρόβλημα χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν θα έχετε το λόγο για δύο λεπτά ο καθένας. Κάθε συντονιστής από δύο λεπτά. Η κυρία Μέτσολα. Είναι στην αίθουσα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε το πάνελ που μας συνάντησε σήμερα και μας ενημέρωσε για τα όσα συμβαίνουν ε, ε, για τη, όσα γίνονται στις χώρες που αντιμετωπίζετε, κυρίως ε, τα εγκατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι σύμπτωμα της όλης συζήτησης φυσικά, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στιγμή για ψυχραιμία ε, και να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις, διότι όπως είπαν και οι υπουργοί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ε, τη μεταναστευτική κρίση, αλλά και μια πάρα πολύ σημαντική κρίση υγείας. Όσον αφορά την Τουρκία, δεν μπορούμε να της επιτρέπουμε να εκβιάζει και πάλι την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τους πιο ευάλωτους ανθρώπους του πλανήτη ως πιόνια σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι ισχύω. Είναι απαράδεκτο και είναι και ανεύθυνο. Ταυτόχρονα ακούσαμε από τους Έλληνες υπουργού, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι δίνεται πολύ βοήθεια στην Ελλάδα, ε, ότι υπάρχει αλληλεγγύη ε, και νομίζω ότι σε τέτοιους ευάλωτους καιρούς είναι πάρα πολύ σημαντικό οι χώρες στην πρώτη γραμμή ε, που αντιμετωπίζουν τόσο επίγοντα ζητήματα να βρίσκουν βοήθεια από μια Ευρώπη ενωμένη που μπορεί να επιδείξει αλληλεγγύη. Ε, πέραν ε, το πιο μακρυπρόθεσμων ε, θεμάτων, την μεταρρύθμιση του Διβλίνου και ενό νέου συμφώνου για τη μετανάστευση που πρέπει να τα συζητήσουμε στη διάρκεια αυτή τη θητεία, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και τα πιο επίγοντα ζητήματα τα οποία θα αναπτύξω τώρα. Καταρχά, προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσατε να μου πείτε λίγο περισσότερα για του διάβλου επικοινωνία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα με την Τουρκία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη εχθέ με την Κριστιάνα Μαμπούρ να λέει ότι ότι δεν έχουν υπάρξει περισταστικά ε, μετάδοσης στο νησί ακόμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για ένα τέτοιο σενάριο. Ε, η Επιτροπή δεσμεύεται να αναθεωρεί την κατάσταση περιοδικά στην Ελλάδα και να προσαρμόσει Ελπίζω να πέρασε η τελευταία ερώτηση. Δυστυχώ όχι, χάθηκε το μικρόφωνο τη ομιλήτρια. Όσον αφορά τι δεσμεύσει ε, που ανέφερε η Επίτροπο Γιώχανσε για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορείτε να μα πείτε κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε για το χρονοδιάγραμμα η κρίση υγείας, η πανδημία αυτή ε, καθυστερεί ή δεν επιτρέπει τη μετεγκατάσταση αυτών των ε, ανηλίκων. Ε, ωραίες και καλές οι δεσμεύσεις, αλλά πότε θα ξεκινήσουν ε, οι μετεγκαταστάσεις. Και τέλος, είδαμε σε μία επιστολή που ε, μας έστειλαν ο Αντιπρόεδρος Κοινάς και Επίτροπος Γιώχανσαν ε, τα 250 ευρώ τα οποία δεσμεύουμε για τη διαχείριση των προσφάτων αφήξεων από την Τουρκία. Λίγο περισσότερα ε, στοιχεία. Τι γίνεται με υγειονομικέ εγκαταστάσεις, ε, δίνονται χρήματα εκεί ή θα πρέπει η Ελλάδα να πληρώσει το λογαριασμό μόνη τη. Και τέλος, όταν αναφερόμαστε σε τέτοια συνδρομή, θα ήθελα να ακούσω και ε, τα όσα θα μας πει η Frontex. Ε, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η πανδημία σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο προσωπικό επιτόπου για να παράσχει βοήθεια. Ε, ναι, μεν δίνουμε χρήματα, αλλά έχουμε δει ότι υπάρχει ανάγκη για επιπλέον προσωπικό επιτόπου. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μία εικόνα ε, του τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, είστε εδώ, μ' ακούτε. Μπορείτε να λάβετε το λόγο. Έχετε δύο λεπτά. Ναι, ωραία, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που ακούσαμε μέχρι στιγμής. Πολλοί ανέφεραν την ανάγκη αλληλεγγύης και νομίζω πως ε, τώρα που είδαμε μονομενες αποφάσεις των κρατών μελών στην υγειονομική κρίση είδαμε ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνο του. Αυτό ισχύει για τη μετανάστευση, την οικονομία, την υγεία. Απαιτείται λοιπόν πραγματική αλληλεγγύη. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, αυτό δεν το βλέπω από όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σχοινά, τον αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, πώ χρησιμοποιεί ακριβώ την αρμοδιότητά του ω Αντιπρόεδρο τη Κομισιόν για να πιέσει τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει και άλλες ε, μόνο από κοινού πώς θα επανέλθει η αλληλεγγύη και η συνεργασία. Η Επίτροπος Γιώχανσον μίλησε ε, για το ότι υπάρχει μια διαφορά. Τώρα προσπαθούμε να περάσουμε σε μια αποσυμφόρηση των δομών. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει γρήγορα για να μην έχουμε κορονοϊό στα νησιά. Θα μπορούσατε ίσως εσείς ή οι Υπουργοί ε, να μας πούν πού βρισκόμαστε όσον αφορά την ε, έβρεση θέσεων σε σπίτια ή ξενοδοχεία, πόσες θέσεις έχουμε και πόσα κράτη-μέλη μέχρι στιγμή συμμετέχουν στην μετεγκατάσταση ασυνόδευτών ανηλίκων και μήπως αυτά τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ε, να δεχτούν και οικογένειες και να δουν την επανένωση των οικογενειών. Θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση προς την κυρία Γιώχανσον αλλά και στους υπουργούς ε, στην Ελλάδα τι ε, εννοούν τώρα με τις ε, δομές, μιλήσατε για νέες δομές, ε, θετικό αυτό, αλλά αντιλαμβάνουμε ότι είναι κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Θα ήθελε να γνωρίζω πώς θα οργανωθούν, θα είναι ανοιχτά ή κλειστά, για πόσα άτομα και υπάρχουν ε, όχι μόνο τα λεφτά αλλά και το προσωπικό εκ των προτέρων για να οργανωθούν. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα σταματήσω εδώ για να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο μας με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Ινετφέλντ από το Renew Europe. Μας ακούτε. Μπορείτε να μιλήσετε. Κυρία Νιτφέλντ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. We will continue with... Θα συνεχίσουμε ε, την κυρία Ταντίνο από το ID. Α, όχι, ο κύριος Λετζέρη. Έχετε τον λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με ακούτε. Ναι, κάθαρα. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που με προσκαλέσατε και οργανώσατε αυτήν την συνεδρίαση υπό αυτές τις συνθήκες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω από τη σκοπιά της Frontex για την κατάσταση στα ελληνικά σύνορα. Πρώτα απ' όλα να σου πω τι συμβαίνει. Και κόβεται η μετάδοση. Bon. Ε, Μάλιστα. Κυρία Ινετφέλντ, με ακούτε. Έχει τον λόγο. Ναι, ναι, σε μένα μιλάτε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ε, ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα στον Επίτροπο, στην Επίτροπο Γιώχανσον. Το έχουμε ξαναπεί για την ε, εκένωση, επαναγκατάσταση ανθρώπων που είναι, έχουν κολλήσει στα νησιά. με διάφορα ονόματα χωρών και αριθμών. Μπορείτε να μας δώσετε έναν οριστικό κατάλογο ποιες χώρες έχουν δεσμευτεί ότι θα με αντικαταστήσουν άτομα, ποιες θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι σημαντικό για να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Δεύτερον, τι κάνει η Κομισιόν για τις χώρες πλην Ελλάδος ε, που ανέστηλαν το δικαίωμα ασύλου, που απλά καταγράφουν ανθρώπους, αφήξει αφήξεις δηλαδή. Μετά οι αφήξεις από 1η Μαρτίου στην Ελλάδα ε, καταγράφονται μόνο από την αστυνομία και την Frontex και κρατούνται σε άσχημες συνθήκες. Θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις γιατί ε, ακόμα και αν ανασταλεί το δικαίωμα ασύλου, δικαίως ή όχι, νομίζω η μεταχείριση που λαμβάνουν από την αστυνομία και την ε, Frontex, ε, όχι δηλαδή τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι πολύ ενισχυτική. Τέλος, προς τον κύριο Λετζέρη που θα μιλήσει αμέσως μετά και θα μπορούσε να απαντήσει. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να γνωρίζω θα ερευνήσετε πλήρως και ε, θα μας ενημερώσετε για όλα αυτά τα οποία ακούγονται για δυσανάλογη βία και αποθήσεις παραδείγματος χάρη να ακούσαμε ότι κάποιοι δανείοι της Frontex αρνήθηκαν να εκτελέσουν ε, διαταγή για απόθεση και μετά ακούσαμε κάποιες φήμες ότι τα κράτη-μέλη σκέφτονται να αποσύρουν ε, τις ε, δυνάμεις τους ε, από την Frontex, από τα ελληνικά σύνορα, λόγω COVID, λόγω του ιού. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί αν αρχίσουν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους τα κράτη-μέλη έχουμε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ένετφελτ, κύριε Λετζέρη. Ναι, ακούτε. Κύριε Λετζέρη. Πιέστε το κουμπί παρακαλώ. Ναι, περιμένουμε. Ωραία, συνεχίζουμε με την κυρία Ταρίνο από το ID. Με ακούτε? Με ακούτε κύριε Ταρίνο. Όχι. Συνεχίζουμε με την κυρία Στρίκα τους πράσινους. Κυρία Στρίκ, με ακούτε. Όχι. Α, ναι, έχετε τον λόγο. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές ε, της ακρόασης αυτές. Καταρχάς να τονίσω ότι ήδη αντιμετωπίσαμε ανθρωπιστική κρίση λόγω της, ε, του υπερπληθισμού των ελληνικών νησιών. Οι μετανάστες ε, ε, ήταν μόνοι τους και υπήρχε έλλειψη όλων των βασικών αναγκών για όλους. Αυτό ακριβώς ε, μετατράπηκε σε μια κατεπίγουσα κρίση υγείας γιατί δεν υπάρχουν υγειονομικοί χώροι, δεν υπάρχει χώρος απομόνησης και το καθεξής. Αν δω τα μέτρα αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί πριν από την κρίση του κορονοϊού. Αν δείτε τα εκατομμύρια στον προπολογισμό θα δείτε ότι τα 50 εκατομμύρια και μόνον δίνονται για ιατρική περίθαλψη. Ε, νομίζω ότι αυτά δεν είναι επαρκή. Η μετεγκατάσταση είναι περιορισμένη μόνο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και μάλιστα 1.600 και μόνο από αυτούς, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε προληπτική εκένωση όλων των ευάλωτων του Ντονάσολο από τα νησιά, καθόν επίσης και πολλοί γιατροί ζήτησαν να υπάρχει προληπτική εκένωση και ε, είπαν ότι η προστασία ε, κατά του ιού και ενώ ταυτόχρονα θα παραμένουν στο νησί δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό γιατί δεν υπάρχει χώρο για κάτι τέτοιο. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει χώρο στην ενδοχώρα για να γίνει αυτή η εκένωση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σίγουρα πολύ περισσότερε δυνατότητε στην ενδοχώρα. Τι γίνεται με διαθέσιμη στέγαση, ξενοδοχεία, όπω έχει γίνει κάποια έρευνα και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πιέσει, να ζητήσει, ε, να εκενωθούν τα νησιά. Επίση, επίσης, το Συμβούλιο. Τι κάνει το Συμβούλιο για να πιέσει τα κράτη-μέλη για περισσότερη μετεγκατάσταση και ε, σε άλλες κατηγορίες, όχι μόνο τους μία συνόδευτούς ανηλίκους και ε, για να υπάρχει και ε, γρήγορη επανένωση οικογενειών και να προχωρήσουν και αυτές οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει πρόσφαση σε νομική συνδρομή και ανθρωπιστική βοήθεια και φυσικά αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτή τη στιγμή δεδομένων των συνθηκών αλλά και για τις νέες αφήξεις ε, πιο συγκεκριμένα. Η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφαγες δεν έχει πρόσβαση. Τι γίνεται για αυτές τις, τους ισχυρισμούς για επαναπρόθεση στα νησιά, pushbacks και τι γίνεται και για τι δεσμεύσει ε, για τι αιτήσει ασύλου. Ε, Μήπω μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι, αφού ξεκινούν και πάλι οι διαδικασίε ε, υποδοχής αιτήσεων ασύλου, θα θέλαμε κάποιε περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες. Έχει υπάρξει ε, Όντω, μη επέλαση θα, ήθελα να, απέλαση, θα ήθελα να ζητήσω να μην υπάρχει κράτηση και απέλαση όταν η τουρκική κυβέρνηση δεν δέχεται καμία επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Στρίκ. Ο κύριος Λεζερή. Με ακούτε, κύριε Λεζερή. Όχι. Συνεχίζουμε με την κυρία Ταρίνο από το ID. Μπορείτε να με ακούσετε. We wait for you. Κυρία Ταρντίνο, περιμένουμε. Please Παρακαλώ, πατήστε το κουμπί. Μπορείτε να μιλήσετε. Κυρία Ταρντίνο. Yes. for one minute. Περιμένουμε ένα λεπτό. Push the button, Mrs. Tardino. Κυρία Ταρντίνο, πατήστε το κουμπί. Α, χάθηκε πάλι. Πάμε πάλι, παρακαλώ. Πιέστε το κουμπί. Κυρία Ταρντίνο, έχετε το λόγο. Πάλι, πατήστε πάλι. Twice. Once. Yes. Um, Mrs. please. Κυρία Ταρντίνο, παρακαλώ. Πιέστε σας παρακαλώ το κουμπί. Okay. Oh. Une fois et attendre. Okay. Which ones? And Πατήστε και περιμένετε. Πατήστε το κουμπί και περιμένετε. Έχετε το λόγο. Α, α, να τη. The micro doesn't work. Doesn't work. Oh, we continue with. Συνεχίζουμε με τον κύριο Προκατσίνη από το ECR. Με ακούτε, κύριε Προκατσίνη. Mr. Procaccino. Κύριε Προκατσίνο. Έχετε το λόγο. Πατήστε το κουμπί, παρακαλώ. Δεν ακούγεστε. doesn't work. Okay, can you refresh the page? Ε, ανανέωση στη σελίδα, κύριε Προκατσίνου. Μ' ακούτε τώρα? Ωραία. Καλημέρα, με ακούτε? Τέλεια. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές που έλαβαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τις ελληνικές αρχές ιδιαιτέρως για την πολύ σκληρή δουλειά που κάνουν σε αυτή την κρίση η οποία επιδεινώθηκε από την ε, κατάσταση σε υγειονομικό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι σωστά όλα τα μέτρα οικονομικής ε, βοήθησης και βοήθειας και επιχειρησιακής βοήθειας προς την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ επίσης ότι είναι δίκαιο και απαραίτητο να ασχοληθούμε με την κατάσταση ε, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Αλλά ανησυχώ ιδιαίτερα, ακούγοντας και κάποιους συναδέλφους, ε, με την περίπτωση να εκμεταλλευτούμε αυτή την ε, υγειονομική κατεπίγουσα ανάγκη για την ε, μετεγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι είναι παράδοξο δεδομένου ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση, δεν μου επιτρέπεται να πάω ούτε καν στη διπλανή πόλη ε, από αυτή που διαμένω. Ε, και να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να κατανείμουμε δεκάδες χιλιάδες ε, παράτυπους μετανάστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτηκα είναι το κλασικό ε, ο κλασικός δούριος ύπος, ε, να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την ε, κατάσταση της υγειονομικής κατεπίγουσας ανάγκης για να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα δημόσιας τάξεως στην Ευρώπη και ε, υγειονομικής τάξεως σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ θεωρούμε ότι είναι η στιγμή να υπάρξει μια πολύ ισχυρή δράση αντιμετώπισης ε, των αναχωρήσεων ε, των ε, παράτυπων μεταναστών, διότι το να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα Άμα τη αφήξη του στην Ευρώπη ε, σε ένα ε, ελληνικό νησί, για παράδειγμα, είναι κάτι το παράλογο. Ε. Είναι ένας παραλογισμός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και περαιτέρω προβλήματα σε οικονομικό επίπεδο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις χώρες καταγωγής τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ να έχουμε την κοινή λογική, τον κοινό νου, να σκεφτούμε και την ε, κατεπίγουσα ανάγκη λόγω υγείας και το πώς να μην επιδεινώσουμε αυτή την, αυτή την κατεπίγουσα ανάγκη. Και όσον αφορά και τη σχέση με την Τουρκία, θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε ένα επιπλέον παράδοξο. Το να θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε προσοχή και να ρίχνουμε χρήματα στον ε, Τούρκο πρόεδρο ε- Ερντογάν σημαίνει ότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας ότι η Ευρώπη θα πρέπει κυρίως να δείξει αλληλεγγύη στην Ευρώπη, στις χώρες της όπως την Ελλάδα και να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τις χώρες αυτές από εξωτερικές επιθέσεις. Εγώ δεν έχω να θέσω ερωτήσεις ε, στους Έλληνες υπουργούς. Θα ήθελα απλώ να τους ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Ελλάδα για τη δουλειά που κάνει, διότι ε, Καθώς υπερασπίζεται τον ελληνικό λαό, υπερασπίζεται τους λαούς όλης της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ταρντίνο από το ID. Με ακούτε? Μπορείτε να μιλήσετε, να πατήσετε το κουμπί. No. We will continue. Ωραία, θα συνεχίσουμε με την κυρία Έρνστ. Η κυρία Έρνστ από την ΚΟΕ. Είστε εδώ κυρία Έρνστ. No. We wait for a minute.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 Mr. López Aguilar, our Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ, ο πρόεδρος μας. Με ακούτε? Mr. López Aguilar. Κύριε Λόπεθ Αγγιλάρ, με ακούτε? Κύριε Πρόεδρε. No. We wait. Okay. Oh. Chair. Hello. Okay. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και σας ευχαριστώ που πραγματικά ανταποκρίνεσαι στις δεσμεύσεις της Επιτροπής μας παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τις συνθήκες. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους και βεβαίως συμφωνώ και εγώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα θέματα και να κάνω τρία ερωτήματα, δύο προς την Κομισιόν και ένα προς τους ε, υπουργούς, ε, τις ελληνικές αρχές ε, που μας αφιερώνουν το χρόνο τους. Πρώτα προς την Κομισιόν. Πότε θα γίνουν αυτά αυτά, αυτοί οι 1600 ασυνόδευτοι ανηλικοί θα μεταφερθούν πρώτα στην υπηρετική Ελλάδα και μετά στις χώρες εκείνες που δεν έχουν ακόμα κατανομαστεί, που είναι διατεθειμένες να τους μοιραστούν. για να έχουμε αυτή την πρώτη ε, πρωτοβουλία με ε, Η άλλη ερώτηση απευθύνεται προ την Κομισιόν. Τα 350 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναφέρθηκαν ε, να διατεθούν για τον ε, σκοπό ακριβώς που πρέπει, πώς ε, θα το διασφαλιστεί. Γιατί έχουμε ακούσει μαρτυρίες ότι κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, κληρώσει τον στόχο τους γιατί έχουν υπάρξει ε, κάποιες ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες και τελικά δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Και η τρίτη ερώτηση απευθύνεται προς τις ελληνικές αρχές. Ποιο είναι το σχέδιο ανάγκης εάν υπάρξει κάποια έξαρση του ιού στις δομές στις δομές που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής αλλά είχαμε ε, κρούσματα στα νησιά που βρίσκονται οι δομές. Τι θα γίνει αν υπάρξουν ε, τέτοια κρούσματα. Θα είναι περιορισμένοι εκεί οι άνθρωποι χωρίς ιατρική περίθαλψη, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες. Ε, θα έχουμε θανάτους επιτόπου. Ποιο είναι το σχέδιο ανάγκης ποια είναι τα μέτρα για να αποσυμφορηθούν οι δομές αυτές για να υπάρξουν μετεγκαταστάσεις σε ασφαλή μέρη ε, για τα πιο ευπαθή άτομα. Τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις δηλαδή για να εκμεταλλευτώ τον χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Νταλή είναι εδώ. Ε, συντονιστής της ΓΚΟΕ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ομιλητές. Οφείλω να πω ότι όλα αυτά είναι κάπως μονομερή. Ακούσαμε διασφάλιση των συνόρων της Ευρώπης, αλλά δεν ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για τις υποχρεώσεις που υπάρχουν για διασφάλιση των θεμελιωτών δικαιωμάτων και υπάρχουν κάποια ζητήματα και προ της κρίσης του ιού. Και ο Υπουργό είχε έρθει τον Νοέμβριο, μας είχε πει ότι υπάρχουν χιλιάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι. Επ' αυτού λοιπόν του ζητήματος θα ήθελα να γνωρίζω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά έχω και κάποια άλλα ερωτήματα στα οποία θα ήθελα να εστιάσω. Όσον αφορά τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Μηταράκη, ε, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστήριων επισκέφθηκε την Ελλάδα πριν από 15 μέρες και υπάρχουν κάποια πρόωρα ευρήματα με άμεσα μέτρα που ζητούν να ληφθούν για την κατάσταση στα νησιά. Ποια ήταν αυτά τα μέτρα και τι έχουν κάνει οι ε, ελληνικές αρχές. Μπορείτε να δημοσιεύσετε αυτήν την έκθεση και Σα ερωτώ, θα την δημοσιεύσετε. Κυρία Γιωχάνσεν, κυρία Επιτροπέ, ε, θα ήθελα να γνωρίζω αν ε, έχετε ζητήσει αυτή την έκθεση από τις ελληνικές αρχές, αν όχι γιατί όχι, δεδομένου του ότι το δικό σας το τμήμα είναι υπεύθυνο για εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ ε, των Ευρωπαίων φορολογουμένων που πηγαίνουν για να χρηματοδοτήσουν δομέ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια βήματα έχει κάνει η κυρία Ιωχάνσεν. Γιατί δεν ασκήσατε κριτική στο προεδρικό διάταγμα που ε, προέβλεπε προσωρινή άρση του δικαιώματος υποβολής αιτήματο ασύλου τον Μάρτιο, το οποίο βεβαίω τώρα εξέπνευσε. Αλλά τι ε, γίνεται, τι έχετε κάνει εσείς ακριβώς για τις παραβιάσεις αυτές του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα γνωρίζετε και θα ήθελα να σχολιάσετε τις εκθέσεις στα ελληνικά ΜΜΕ ότι ένα νέο νόμο περί μετανάστευση συντάσσεται από το αρμόδιο Υπουργείο, ο οποίο παραβιάζει κατάφορα το ευρωπαϊκό δίκαιο, προτείνει οι αιτούντε άσυλο να μην έχουν την επιλογή ε, προσωπικής συνέντευξης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη η γλώσσα, αν έχουν μείνει σε άλλη χώρα πάνω από δύο μήνε ε, όπου δεν απειλούνται η αίτησή τους ε, δεν θα γίνεται δεκτή. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Και τέλο για ε, να επανέλθω ε, στους Έλληνες υπουργούς. Ενημερώθηκε τώρα μόλις ότι στην δομή της Σύρου ε, υπάρχουν, υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την ασφάλεια. Γιατί δεν το κάνει η αστυνομία. Θα επαναληφθεί αυτό στο μέλλον. Και τι γίνεται ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χέρμστ αντιπρόεδρος τη Επιτροπής Προϋπολογισμού. Με ακούτε. Herbst. Κύριε Χέρμπστ, παρακαλώ, με ακούτε. Με ακούτε, ωραία. Ευχαριστώ, ωραία τότε. Ωραία, εξαιρετικά. Να πω δύο λόγια εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να αναφερθώ στο σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού, το οποίο προτάθηκε πριν από λίγες ημέρες, που είναι και το πιο σημαντικό θέμα για μας, για την κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σα διαβεβαιώ ότι εμεί στην Επιτροπή Προπολογισμών έχουμε στόχο να ε, προχωρήσουμε την πρόταση αυτή το συντομότερο δυνατόν. Ε, γνωρίζετε ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Ε, δεν ξέρω ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ημέρες, αλλά πραγματικά θέλουμε να προχωρήσουμε το, το δυνατόν πιο γρήγορα. Εξαρτώμαστε βεβαίω και από το Συμβούλιο, θα πρέπει να το έχετε και κατανό αυτό. Είναι ο άλλο βραχίωνα τη ε, αρχή προπολογισμού και θα πρέπει ίσω να ε, ε, πιέσουμε και αυτού ίσω. Και επειδή η Επίτροπο Γιώχανσον ήδη σα είπε ποια είναι αυτά τα επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ και πού θα διαπανηθούν, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το συνολικό επίπεδο χρηματοδότηση του παρόντο πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου ήταν πάρα πολύ χαμηλό και ότι ο Εθνικό Φάκελο για την Ελλάδα για το θέμα αυτό ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Ε, πρέπει λοιπόν να αντλούμε και εμεί διδάγματα από το ε, λάθη μας, ε, διότι δεν ήμασταν αρκετά ευέλικτοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι συνθήκε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στι συζητήσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα γίνουν τις επόμενε εβδομάδες. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι ε, για ένα πιο φιλόδοξο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και νομίζω ότι οι υπηρεσίες, ε, θα συμφωνήσει και ο Frontex εδώ, θα πρέπει να έχουν ένα φιλόδοξο πι ώστε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την κυρία Ταρντίνο. Με ακούτε τώρα? Κυρία Ταρντίνο, παρακαλώ. Πατήστε το κουμπί. Περιμένουμε ένα λεπτό. Ναι. Όχι. Πάμε πάλι κύριε Ταρντίνο. Ναι. Όχι. Ε, θα τα καταφέρετε κύριε Ταρντίνο. Δοκιμάστε ξανά κυρία Ταρντίνο. Um, uh, κυρία Ταρντίνο, ε, θα μιλήσει τηλεφωνικά. Ο κύριος Λεζερή θα μιλήσει τηλεφωνικά θα μιλήσει μέσω κινητού τηλεφώνου. You have the floor, Mr. Legeri. Έχετε το λόγο, κύριε Λεζερή, για 7 λεπτά. Αυτό δυστυχώς δεν μεταφράζεται. Uh, honorable members of the parliament, distinguished participants, thank you for the invitation uh, and I will uh, present from project perspective the situation at the Greek border. At the beginning of March, we got a request from Greek authorities to launch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

One ευχαριστώ. Μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Τα μέλη που δεν μπόρεσαν να λάβουν το, γνώμο, το λόγο σήμερα μπορούν να στείλουν ερωτήσεις ε, στην ε, γραμματεία της ε, Επιτροπής που θα τα διαβιβάσει στου ομιλητέ για να απαντήσουν γραπτώ. Και θα προσπαθήσουμε τέλος να μιλήσουμε με την κυρία Ταρντίνο. Με ακούτε? Κυρία Ταρντίνο. Μπορείτε να προσπαθήσετε. Όχι. Περιμένουμε ένα λεπτό. Κυρία Ταρντίνο, πιέστε το κουμπί. Όχι, δεν λειτουργεί. Ωραία. Περνάμε πάλι στους ομιλητές μας για να ακούσουμε τις απαντήσεις. Ξεκινούμε με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Με ακούτε? Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Τις απαντήσεις σας, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Σύντομα θα απαντήσω σε ε, δύο ζητήματα. Το ένα αφορά, ακούστηκε μία παρατήρηση σε σχέση με pushback, με αποθήσεις και θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις φήμες που κυκλοφόρησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γίναμε αποδέκτες fake news τα οποία αποδείχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες πόσο παραπλανητικά ήταν, σας θυμίζω ότι ο κύριος Ερντογάν την πρώτη μέρα είπε ότι 60.000 ήδη οδεύουν προς Ευρώπη. Και την επόμενη μέρα είπε ότι έχουν φτάσει τις 160.000. Ε, λέγοντας ουσιαστικά ψέματα για να διαμορφώσουν ένα κλίμα προκειμένου να οθήσουν και άλλους ανθρώπους δυστυχισμένους να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν την ελληνοτουρκική μεθόριο. Θέλω να σας πω λοιπόν με κάθε εντυμότητα και ειλικρίνεια ότι ό,τι έγινε όλες αυτές τις μέρες στην ελληνοτουρκική μεθόριο έγινε υπό το φως δεκάδων ή εκατοντάδων μέσων ενημέρωσης από όλο τον κόσμο. Θέλω να πω ήταν πάνω από 50 ε, κανάλια στην περιοχή και ειδησιογραφικά πρακτορία και όταν ένα πράγμα, ένα γεγονός το καταγράφουν χιλιάδες μάτια και το ακούνε χιλιάδες αυτιά, δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Και δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα. Όλα έγιναν υπό το φως της ημέρας της δημοσιότητας. Μα κυρίως την ώρα που οι ελληνικές δυνάμεις, όπως σας είπα, δέχονταν επιθέσεις για τις οποίες κινδύνευε η ζωή τους αντέδρασαν με ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Είμαστε στην ίδια γραμμή. Είμαστε με τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, είμαστε με τις αξίες του ευρωπαϊκού δικαίου ασύλου, είμαστε μαζί στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστατεύουμε στην πράξη καθημερινά την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στις ε, πανανθρώπινες αξίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που θέλω να σας παράσχω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και αυτό θα κάνουμε παρά την τεράστια πίεση που όλοι αναγνωρίζετε δέχεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε σχέση με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να ε, τονίσω έχει να κάνει με τη Frontex. Θέλω να σας πω ότι σταδιακά και σε συνεννόηση στη συνέχεια με τον κύριο Λεζερή ε, κάποιες δυνάμεις θα αποχωρήσουν, κυρίως αυτές σε πρώτη φάση που ήρθαν με μια διμερή συμφωνία και θέλω και πάλι να τις ευχαριστήσω. Ε, τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που λαμβάνονται για το προσωπικό και της Frontex αλλά και των ελληνικών αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων είναι πάρα πολύ αυστηρά και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε αυτά τα μέτρα γιατί αυτό που κυρίως προέχει αυτή τη στιγμή είναι για να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα, για να κρατήσουμε όρθια την Ευρώπη, τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία παίζει πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του, της επιδημίας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you. One additional remark. Three minutes each speaker maximum. If need... Μια επιπλέον παρατήρηση, τρία λεπτά ο κάθε ομιλητή. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να στείλετε επιπλέον ε, γραπτές απαντήσεις. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Σχοινά. Είστε εδώ κύριε Σχοινά. Κυρία Γιώχανσον. Ο κύριος Οφλάχερτη. Ναι, παρακαλώ. Τρία λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, ε, διότι ε, δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για μένα, αλλά ε, όσον αφορά τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ε, τη σημασία της εξατομήκευσης για τις αιτήσει ασύλου. Πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει εξατομικευμένη διεκπαιρέωση της άτοσης ασύλου. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στη διάσταση μια κατάσταση που έλαβε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα το πρωί. Την ιδιαίτερη κατάσταση των 2.000 περίπου ατόμων που έφτασαν στη διάρκεια του μηνός Μαρτίου. Μπορεί πράγματι ε, ελάχιστοι από αυτούς να δικαιούνται διεθνή προστασία, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διαδικασίες ε, και να είναι κατάλληλα προβεβλημένες ώστε να καθοριστεί το τι καθεστώς δικαιούνται, σε ατομική βάση, να είναι εξατομικευμένες οι διαδικασίες. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει ένας οξύς κίνδυνος ε, στους καταβλισμούς ε, στην Ελλάδα λόγω του COVID-19. Είναι πολύ δύσκολο να ε, σας εξηγήσω την έκταση του κινδύνου. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είμαστε ευάλωτοι και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Και φυσικά σε ένα καταβλισμό βιογκώνονται αυτοί οι παράγοντες κινδύνου σε έναν απίστευτο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει λοιπόν άμεση απάντηση και να χρησιμοποιηθούν και ξενοδοχειακά και άλλα τουριστικά καταλήματα για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο υπουργό ο κύριο Μηταράκη. με ακούει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω απαντώντας ε, στον Πρόεδρο για τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Ε, ναι, φυσικά υπάρχει επεδρικό ε, σχέδιο σε περίπτωση που υπάρχει κρούσμα, να υπάρχει απομόνωση, να υπάρχουν επιπλέον περιοχές καραντίνας στην εγκύτερη περιοχή των καταβλισμών. Αναφερθήκατε στη μεταφορά των ατόμων σε ασφαλείς χώρου. Για να είμαι δεν είμαι βέβαιος τι είναι ε, ο ασφαλή χώρο ε, Προβλέπαμε να κάνουμε κάποιε μετακινήσει από τη Ριτσίνα, Ριτσόνα, από τη Μόρια συγγνώμη, στη Ριτσόνα ε, και τώρα έχουμε κάποια κρούσματα στη Ριτσόνα. Είναι καλή διαχείριση, υπάρχουν εγκαταστάσει, δεν υπάρχουν προβλήματα όπω στη Μόρια και τελικά το κρούσμα εμφανίστηκε εκεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για μαζικέ εκενώσει των καταβλισμών, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στην ενδοχώρα. Είναι περιορισμένο ο αριθμό των ξενοδοχείων, πολύ ευχαρίστω να του εκμεταλλευτούμε, αλλά θα θέλαμε να συζητήσουμε και τη χρηματοδότηση για τις επιπλέον 40.000 κλίνες που θα χρειαστούν, για πόσο καιρό και πού μπορούμε να τις βρούμε. Για να μην ξεχνάμε και το θέμα της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ε, η θέση, αν η θέση είναι ότι θα τροποποιηθεί η συμφωνία ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των ατόμων εκτός ε, της νήσου και να υπάρχει ακόμα δυνατότητα της επιστροφής τους, διότι ε, μπορεί και να είναι λιγότερο από μισή αυτοί οι οποίοι δικαιούνται διεθνού προστασία και θα πρέπει να επιστραφούν, ακολουθώντας βεβαίως ε, τις ε, ε, νόμιμε διαδικασίε, αλλά δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό εάν δεν υπάρξει μια νέα κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Για αυτού που αφήχθησαν εντό του μηνό Μαρτίου. Υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο ετέθη από το Συμβούλιο τη Ευρώπη και πρόσεξα ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις που έκανα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε δυνατότητα αναμονή ε, εν αναμονή και του κορονοϊού και την ε, ξέσπασμα της Τουρκίας. Τις πρώτες λίγες μέρες λοιπόν δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσει που θα θέλαμε και φυσικά χρειαστήκαμε δύο εβδομάδες, ε, δαπανήθηκαν 8 εκατομμύρια και κάναμε έτσι και χρηματοδότηση για να δημιουργήσουμε δύο προσωρινά χώρου στη Μαλακάσα και στις Σέρες. Μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, υπήρχε και η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για να υπάρχει κατάλληλη ιατρική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 βοήθεια προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε μια διπλή κρίση όπως εξελίχθηκε και συνεργαζόμαστε και στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να το επιτύχουμε. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Μία για τα ε, κέντρα πολλαπλών σκοπών. Θέλουμε να γίνεται εκεί η καταγραφή, ε, να υπάρχουν τα γραφεία του, ασόλ, ασύλου, να υπάρχουν ασφαλείς περιοχές για οικογένειες, για συνόδευτους ανηλίκους, ώστε να μην είναι ε, τμήμα του γενικού πληθυσμού. Γι' αυτό ακριβώς και τα αποκαλούμε και κέντρα πολλαπλών σκοπών. Δεν θα περιορίζονται εκεί από τις ε, οδηγίες οι άνθρωποι, θα μπορούν να ε, εισέρχονται και να εξέρχονται. Θα υπάρχουν κανόνες φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό τα κέντρα αυτά να έχουν ε, κανόνες που να συνάδουν και με τις διεθνείς συνθήκες και τις οδηγίες. Ένα τελευταίο στοιχείο για το άσυλο. Εξετάζουμε τη δυνατότητα να ξαναξεκινήσει η διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου μέσω Skype ή μέσω άλλων μορφών, αλλά είχαμε με μια καθυστέρηση περίπου 35.000 αιτήσεων. Αυτό είναι παραπάνω από τις αφήξεις του 2019 και του 2020 και πραγματικά λοιπόν καθυστερούσαμε πάρα πολύ και είχαμε 19.000 περιπτώσεις τις οποίες είχε ολοκληρωθεί η ε, συνέντευξη αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση. Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν αυτό το χρόνο όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για το κοινό στις υπηρεσίες ασύλου για να εκδοθούν οι αποφάσεις για τις συνεντεύξεις οι οποίες έχουν ήδη διεξαχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε Σχοινά, με ακούτε? Κύριε Σχοινά. Commissioner Skinas. Επίτροπε Σχοινά. Επίτροπε Γιωχάνσον, με ακούτε εσείς? No. Yes. We wait. Ναι. Περιμένουμε. One moment. Yes. Ναι, με ακούτε. Με ακούτε. Ωραία. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και με εντυπωσιάζει το ότι τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για την υπομονή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ε, ε, ασυνόδευτη ανήλικη η κυρία Μετσόλα, είναι τη και Λόπες Αγγιλάρ το ρώτησαν αυτό. Λοιπόν, τώρα με τις ε, ελληνικές αρχές, ε, σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές, μεταβαίνουν σε κάποια κέντρα τράνζιτ, οπότε κινούμαστε αρκετά γρήγορα και υπάρχει βεβαίως εκεί πέρα περιορισμός και γίνονται τεστ πριν ε, μετακινηθούν σε κράτη-μέλη. Έχουμε προσφορές για 1.600 από Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία, Κροατία και Ιρλανδία. Συνεργαζόμαστε και με άλλα κράτη-μέλη. Ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα κράτη-μέλη. Οι πρώτοι θα μετακινηθούν αυτή την επόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο. Επίσης, ε, και το ερώτημα αν υπάρχουν καθυστερήσεις. Ε, ναι, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις ε, ε, σε σχέση με την... σχετίζονται με την κατάσταση του εγκλισμού, του lockdown. Υπάρχουν ελάχιστε πτήσεις στην Κροατία οι εγκαταστάσεις που είχαν ετοιμάσει καταστράφηκαν από τον σεισμό. Και αυτό βεβαίω προκαλεί κάποιες καθυστερήσεις. Ε, προχωράμε όμως γρήγορα, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Για την οικογενειακή επανένωση, η κυρία Ζίπελ το ανέφερε πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο κάνουμε από πλευράς ε, κομισιών είναι ότι συντάσσουμε καθητήρες γραμμές προς ε, τα κράτη-μέλη για να συνεχίσουν στο μέτρο του δυνατού ο συνήθως τις διαδικασίες ασύλου και τα λοιπά και την οικογενειακή επανένωση. Ελπίζω λοιπόν να βοηθήσουμε τα καρτεμέλη και η κυρία Σίπελ και η κυρία Στρίκ να ρώτησαν αν υπάρχουν αρκετά δωμάτια ξενοδοχείων και διαμερίσματα. Δεν έχω τους αριθμούς, αλλά συνεργαζόμαστε με την πατερμοστία του ΟΗΕ, ε, η οποία λέει ναι, για να γίνει η ε, μεταγκατάσταση των ευπαθών ε, από τα κέντρα τώρα γιατί είναι επίγον. Κυρία Μετσόλα και κυρία Στρίκ, με ρώτησαν για την υγεία, εάν αυτό καλύπτεται από τα λεφτά, ναι. Πλέονουμε και για παροχές υγείας και ιατρικό εξοπλισμό και πρέπει να πω ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη διευκόλυναν την Ελλάδα με ιατρικό εξοπλισμό με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας που ενεργοποιήθηκε. Οπότε και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Η κυρία Ταλή μου άσκησε κριτική επειδή δεν άσκησα κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Ε, έγινε αυτό, τα είπε και ο κύριος Υπουργός, ε, ότι ακολουθούμε τις αξίες μας ε, και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς ε, συμβάσεις και είχαμε ένα πολύ ειλικρινή διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση και χαίρομαι ιδιαίτερως για το ότι τώρα θα ξαναξεκινήσει η διαδικασία ασύλου για όσου έφτασαν τον Μάρτιο. Επίση η κυρία Νταλή ρώτησε το τι κάνουμε με τις νέες νομοθετικές προτάσεις, όλες οι νέες νομοθετικές προτάσεις όλων των κρατών μελών, όχι μόνο της Ελλάδας, ε, πάντα μελετούνται από τις υπηρεσίες μου. Οπότε, αν υπάρχει κάτι, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με το Κατσουκέο θα το θέσουμε βεβαίως. Όσον αφορά την έκθεση αυτή την οποία αναφέρατε, ε, εξ να αντιλαμβάνομαι δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Ε, έχουμε κάποια πρώτα ευρήματα που έχουν αποσταλεί σε ελληνικές αρχές. Είμαστε όμως σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι κάτω που λαμβάνουμε υπόψη. Ο κ. Λόπες Αγγιλάρ ρώτησε το πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα λεφτά τα οποία δίνουμε θα πηγαίνουν εκεί όπου πρέπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και συνεργαζόμαστε στενά με την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές και με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Υποδερμοσία του ΟΗΕ. Πολύ καλή οργανισμοί με επαγγελματίες επιτόπου. Έχουμε επίσης ε, και 12 άτομα από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών που εργάζονται νυχθημερών στην Αθήνα και στα νησιά σε πολύ στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις ελληνικές αρχές. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά σωστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ. Κύριε Σχοινά. Όχι. Κύριε Φλάχερτη. Κύριε Γκρέσ. Ήθελα απλώ να επανέλθω στην απάντηση της κυρίας ε, Στρίκ ε, προς την Προεδρία για την ε, μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ελλάδα. Τι κάνουμε για να αυξήσουμε τον αριθμό των κρατών μελών. Για το θέμα αυτό θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι έγινε μια πρώτη συζήτηση για την ανάγκη μετεγκατάστασης των ανηλίκων από την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη στο έκτακτο ε, συμβούλιο που έγινε ε, Συμβούλιο Ιστορικών Υποθέσεων που έγινε στις 3 ε, Μαρτίου. Το ξανασυζητήσαμε στις 13 Μαρτίου. Συνεχίζεται η τακτική ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και οι βιντεοδιασκέψεις που γίνονται δύο την φορές την εβδομάδα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίστηκαν σε μία φορά την εβδομάδα. Αλλά το θέμα αυτό είναι μονίμως την ημερήσια διάταξη και το εξετάζουμε όχι μόνο για τον αριθμό των κρατών μελών που θα συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, αλλά η Προεδρία σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και ε, οι συνήθεις διαδικασίες ε, για αυτή τη διαδικασία ε, κατάσταση να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό. Ελπίζω αυτό να απαντάει στην ερώτηση της κυρία Στρίκ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ε, επιπλέον το οποίο μπορεί να επιθυμεί. Ε, από την Προεδρία είμαστε στη διάθεσή τους για να στείλουμε γραπτός απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε Σχοινά, με ακούτε. No. No. We continue. Commissioner Skinas. Κύριε No. Okay. Όχι. Ωραία. Oh, yes. Ο κύριος Ζωνφλάχερτ έχει ήδη απαντήσει. Okay. But I would like to... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, ε, όλους τους ομιλητές και όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη ε, συνεδρίαση με πολύ δύσκολες συνθήκες μέσω βίντεο διασκέψεων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά η συζήτηση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Η επόμενη συνεδρίαση μπορεί να γίνει μέσα Απριλίου. Θα επιβεβαιωθεί η ακριβής ώρα η ε, συνεδρίαση αυτή απέδειξε ότι λειτουργεί το τεχνικό σύστημα. Θα ε, επεκτείνουμε τη διάρκεια της συνεδρίασης για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να μιλήσουν όλα τα μέλη. Ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας και για την κατανόησή σας. Φροντίστε να είστε ασφαλείς και φροντίστε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ.